Przewodniczący! E, witam koleżanki i kolegów. Συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζω και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε. η συνεδρίαση που είχε διακοπεί στις 6 ε, Μαΐου 2010 επαναλαμβάνεται. Έχω πρώτα απ' όλα κάποιες πληροφορίες. Σήμερα για έκτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση εορτάζει την Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας. Πριν ε, από 20 χρόνια η ομοφιλοφιλία διαγράφηκε από τον κατάλογο ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά της ομοφοβίας και αυτό φαίνεται και στη συνθήκη και στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης αυτό το μήνα είχαμε την 60η επέτειο της διακήρυξης ε, Σουμάν στις 8 και 9 Μαΐου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο είχαμε τις ανοιχτές ημέρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κόσμος μπορούσε να δει από κοντά το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω από 33.000 πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Εδώ, σε αυτή την αίθουσα έγινε μια συνεδρίαση με 800 ε, εκπροσώπους ε, των νέων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε μαζί τους εγώ και 11 ευρωβουλευτές συζητήσαμε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτο θέμα, στη, την 3η ε, 11 Μαΐου είχα το προνόμιο να απονείμω το βραβείο νέων του Καρλομάγνου στο Άχεν. πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν η γερμανική, η ιρλανδική και βουλγαρική συμμετοχή αντιστοίχω. Η γερμανική συμμετοχή ήταν μια συνεργασία 21 κρατών μελών και 24 πολυτεχνείων. Ήταν ένα κοινό τεχνικό εγχείρημα. Το δε βραβείο Καρλομάγνου απονομήθηκε δύο μέρες αργότερα στις 13 του μηνός στον ε, Πολωνό Πρωθυπουργό τον Ντόναλτ Τούσκ. Τέταρτη ανακοίνωση, την εβδομάδα που μας πέρασε ήμουν στη Στοκχόλμη σε μια διάσκεψη προέδρων κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόεδροι ή και αντιπρόεδροι των 40 συνολικά κοινοβουλίων ε, ήταν παρόντες. Μιλήσαμε για την ε, μελλοντική συνεργασία για την επερχόμενη Βελγική Προεδρία και μας ε, φιλοξένησαν οι Σουηδοί συνάδελφοι με την βοήθεια των ε, Ισπανών βουλευτών επειδή η Ισπανία αυτή τη στιγμή προεδρεύει στο Συμβούλιο. Επίσης, θα έχουμε κοινέ συνεδριάσεις επιτροπών και μικτές ε, συνεδριάσεις των κοινοβουλίων. Θα ήθελα τώρα να συγχαρώ δύο χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία, που απέκτησαν νέες κυβερνήσεις, οι οποίες ελπίζω να είναι σταθερές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κυβερνήσεις να είναι σταθερές για να λαμβάνονται και οι αποφάσεις γρήγορα. Εμείς βεβαίως είμαστε η πλευρά της κοινοτική μεθόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική για να λαμβάνονται αποτελεσματικά αποφάσεις προς το συμφέρον των πολιτών της Ένωσης. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Τα δε πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα έχετε στη διάθεσή σας. Υπάρχουν σχόλια. Όχι. Οπότε θεωρείτε πως τα πρακτικά εγκρίνονται. Κυρίες και κύριοι. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Μάουρο. Yeah. Mr. Mario Mauro. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα το πρωί στο Αφγανιστάν δύο Ιταλοί στρατιώτε τη στρατιά τη Τωρινέντζ ε, σκοτώθηκαν από μια απόπειρα